ιστορία με την ψηφοφορία. μισή. Τώρα, η δήλωση της Κομισιόν για την ατζέντα της Ντόχα. Η επίτροψη έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σε δύο εβδομάδες θα ξεκινήσει η ένατη πολιτική διάσκεψη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου με μέγιστη σημασία για την Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου και για το πολυμερές ε, εμπορικό σύστημα. Για πρώτη φορά εδώ και χρόνια ε, έχουμε φτάσει πολύ κοντά στην ε, επίτευξη συμφωνίας για πολλά σημεία της αναπτυξιακής ατζέντα. και αν τα μέλη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου καταλήξουν σε συμφωνία, η έκβαση της υπουργικής διάσκεψης θα είναι μια διευκόλυνση για το εμπόριο και μια συμφωνία που θα αποφέρει τεράστιους καρπούς σε όλους τους εμπόρους στον κόσμο Διευκολύνοντα τι τελωνιακέ διαδικασίε, αυξάνοντα τη διαφάνεια, μειώνοντα τη γραφειοκρατία και επιτρέποντα την ε, ταχύτερη διακίνηση των ε, ε, εμπορευμάτων διασυνοριακά. Όλα τα μέλη θα υποφεληθούν από τη συμφωνία αυτή με μεγαλύτερου δικαιούχου στι αναπτυσσόμενε χώρε και κυρίω στι μικρότερε χώρε ή τι χώρε Η συμφωνία θα βοηθήσει τι λιγοτερο αναπτυσσομενε χώρε. η συμφωνια θα βοηθησει τι χώρε αυτέ να βελτιώσουν τη λειτουργία του τελωνιακού του συστήματο και θα βοηθήσει την ε, ραγδαία ανάπτυξη του περιφερειακού ε, εμπορίου και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παρέχει αρρωγή στις χώρες αυτές για να μπορέσουν να εφαρμόσουν καλύτερα τη συμφωνία. Μια συμφωνία για μια εμπορική διευκόλυνση ε, θα συνοδευτεί με κάποια θέματα γεωργικά, αναπτυξιακά, καθώς και ε, θέματα ιδιαίτερη σημασία για τι λιγότερο αναπτυγμένε χώρε. Ήδη έχει επιτευχθεί συμφωνία για τι κατευθυντήριε γραμμέ ό,τι αφορά του ε, προτιμησιακού κανόνε προέλευση που εφαρμόζονται σε εισαγωγέ ε, από λιγότερο αναπτυγμένε χώρε, καθώ και το θέμα τη εξαίρεση των υπηρεσιών. Έτσι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε παρόχους υπηρεσιών από λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και θα συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της αγοράς υπηρεσιών τους. Παρόλο που είναι σχετικά περιορισμένο αυτό το πακέτο δεν είναι ε, ίσονος σημασία, γιατί πέραν των οικονομικών ε, πλεονεκτημάτων του θα έχει και τεράστιο συστημικό αντίκτυπο γιατί θα αποτελέσει το πρώτο βήμα προς την ε, ολοκλήρωση της αναπτυξιακής ατζέντα της ΔΟΧΑ και στους αναπτυξιακούς στόχους ε, του γύρου της ΔΟΧΑ. Αν στεφτεί με επιτυχία αυτή η διάσκεψη, θα ανοίξει ε, την πόρτα για περαιτέρω διαπραγματεύσεις ε, που θα περιλαμβάνουν και τη γεωργία και την πρόσβαση στην αγορά βιομηχανικών αγαθών. Ένα θέμα που θα πρέπει να ε, αναφερθεί σε πολυμερές επίπεδο και επίσης θα επεκταθούμε σε άλλα θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην εντολή της ΔΟΧΑ, αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικά για το εμπόριο. Ένα κεντρικό σημείο της έκβασης θα είναι και ένα πρόγραμμα εργασιών ε, στο οποίο θα με το οποίο θα επανέλθουν στις διαπραγματεύσεις όλα τα μέλη της Παγκόσμια Οργάνωσης Εμπορίου. Πολλά άλλα θέματα θα συζητηθούν και κατά πάσα πιθανότητα θα συμφωνηθούν στην Υπουργική αυτή διάσκεψη. Κεφαλαιόδου σημασία θα είναι η παράταση της συμφωνίας ε, για τις τεχνολογίες πληροφοριών ε, με τις διαπραγματεύσεις που έχουν επαναληφθεί πρόσφατα και που βαίνουν προς μια αίσια έκβαση. Τέλος, δεδομένης της σημασίας αυτής της υπουργικής διάσκεψης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει το γεγονός ότι ε, θα συμμετέχουν στη διάσκεψη αυτή και ευρωβουλευτές ε, στα πλαίσια μιας κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας ε, και της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας και θα, υπάρχει, θα γίνει και μία διάσκεψη, ε, συνέντευξη τύπου με τους ευρωβουλευτές. Σας ευχαριστώ. Τώρα θα δώσω το λόγο στους ομιλητές εκ μέρους των ομάδων. Πρώτα, κύριο Ζάλμπα Μπιντεγκάιν, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστώ για τα λόγια σας. Η διεθνή χαρακτήρα τη οικονομία, η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας θα αποτελέσει αναφυσβήτητα ακρογωνιαίο λίθο τη οικονομικής ανάπτυξης και γι' αυτό χρειαζόμαστε μεγαλύτερη οικονομική απελευθέρωση, λιγότερου τελωνιακού δασμούς και λιγότερου τελωνιακού φραγμούς. Για να μεγιστοποιήσουμε όμως τον αντίκτυπο αυτής της εμπορικής απελευθέρωσης θα πρέπει να εφαρμόσουμε μακροοικονομικές πολιτικές που θα συνάδουν με την πολιτική αυτή. Για παράδειγμα, δημοσιονομική διαφάνεια, διοικητική απλούστευση, αντίστοιχες φορολογικές πολιτικές και επενδύσεις στην παιδεία και στις υποδομές. Για όλα αυτά ε, θα πρέπει να συνοδεύσουμε την πολυμέρεια και τις πολυμερείς συμφωνίες με κάποια πολιτικά μέτρα και μάλιστα η συμφωνία Aid for Trade της Ρώμης, βοήθεια για το εμπόριο του Ιουλίου του 2013, ε, τόνισε τη σημασία αυτής της πτυχής. Βέβαια, πολλά έχουμε ακόμα να επιτελέσουμε, πολύ δρόμο έχουμε ακόμα να διανύσουμε. Συμφωνώ πάντως μαζί σας ότι είναι σημαντικό να, ευκολύνει να ε, λάβουμε υπόψη τους διευκολυντές του εμπορίου, ε, ένας ρόλος πολύ σημαντικός για τις αναπτυσσόμενες χώρες αλλά και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης θα ήθελα να χαιρετήσω την ε, έναρξη της συμφωνίας για τις υπηρεσίες, τη γνωστή ίσα. Είμαι πεπισμένος ότι και αυτή η συμφωνία θα είναι μοχλός ανάπτυξης για τις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά και για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες προκειμένου να βελτιώσουν ε, την ανταγωνιστικότητά τους. Το ίδιο ισχύει και για τις αναπτυγμένες χώρες. Είναι πολύ σημαντική η δέσμευση και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ολόκληρη τη Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ και ευχαριστώ την κυρία Επίτροπο. Σα ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στον κύριο Μορέιρα για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Όπως και στο παρελθόν, πριν τις ε, υπουργικέ διασκέψεις Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου, η Επιτροπή ε, του Διεθνούς Εμπορίου υιοθέτησε ψήφισμα για την παρούσα κατάσταση της αναπτυξιακής ατζέντας της Δόχα και τις προπαρασκευαστικές ε, ενέργειες εν ώψη της υπουργική Διάσκεψης της ΠΟΗ. Το ψήφισμα αυτό της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου θα ψηφιστεί την 5η στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως είπατε, οργανώνουμε και κοινοβουλευτική διάσκεψη. Ε, συνδιοργανώνουμε μάλιστα μαζί με την Διακοινοβουλευτική Ένωση μια τέτοια κοινοβουλευτική διάσκεψη, γιατί μια ισχυρή κοινοβουλευτική διάσταση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου θα αποφύγει την διάβρωση του διεθνούς εμπορίου και θα εξασφαλίσει τη διαφάνεια και νομοποίηση στην Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου. 3 ε, ε, με 6 Δεκεμβρίου θα γίνει στην Ινδονησία ε, η υπουργική αυτή διάσκεψη και περιμένουμε με ανυπομονησία μια αίσια έκβαση αυτής της υπουργικής διάσκεψης. επιταχύθηκαν οι προπαρασκευαστικές ενέργειες από τις αρχές Σεπτεμβρίου υπό την ηγεσία του νέου ε, Γενικού Διευθυντή του, της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου, του κ. Αζεβέντο. Ε, και φυσικά έχουν αντατικοποιηθεί αυτές οι προετοιμασίες τις τελευταίες εβδομάδες. Το αποτέλεσμα βέβαια είναι αβέβαιο ακόμη, αλλά ευελπιστούμε ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία στα βασικά θέματα των διαπραγματεύσεων που είναι η γεωργία, το εμπόριο, η ανάπτυξη, η διευκόλυνση του εμπορίου, που όπως ε, επισημάνετε κι εσείς είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία του πακέτου που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση. Πάνω απ' όλα όμως θα πρέπει να αναζωογονήσουμε και τον διαπραγματευτικό αλλά και κανονιστικό πυλώνα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου. Μία αποτυχία αυτή τη στιγμή θα ήταν εξαιρετικά επιζήμια για το κύρος ε, και ε, τη φήμη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου. Ευχαριστώ κύριε Σερινάλτη. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, παρακολουθούμε με προσοχή τι διαπραγματεύσει που είναι εξελίξει στη Γενέβη ε, με πολύ εντατικό ρυθμό. Είμαστε δίπλα στην Κομισιόν, η οποία ακόμα μια φορά δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πιο ε, ενδιαφερόμενη δύναμη για να δώσει ε, νέα όθεση σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, γιατί ο πλούτος δεν κατανέμεται ε, σωστά. Ε, πρέπει να έχουμε καλύτερες ευκαιρίες για τις αντισόμενες χώρες. Έχουμε πολλές προσδοκίες για τη διευκόλυνση για το εμπόριο, ε, μείωση της γραφειοκρατίας, Δυνατότητε με, μεγαλύτερες για τις μικρομεσαίες μα επιχειρήσει να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην παγκόσμια αγορά. Φυσικά παρατηρούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν γίνεται λόγος για διαφθορά, δεν μιλάει κανένας για φορολογική δικαιοσύνη, δεν υπάρχουν αυτές οι λέξεις στα προπαρασκευαστικά έγγραφα. Ε, αυτά τα θέματα τα αριθμίζουν οι εθνικέ νομοθεσίε, Ελπίζω όμω η Ευρωπαϊκή Ένωση να, ακού, να διατρανώσει τη φωνή της και για αυτά τα θέματα μέσω μιας έστω μονομερούς δικής της θέσης. Δύο ερωτήματα προς την Κομισιόν. Καταρχάς, ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την επικύρωση των δεχομένων συμφωνιών που θα προκύψουν από την Υπουργική Διάσκεψη. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό τόσο σε ό,τι αφορά την ε, Συμφωνία για την Διευκόλυνση του Εμπορίου, την ε, τροποποίηση του ΓΚΑΤΣ για την ε, γεωργική πολιτική, το πακέτο ενισχύσεων για τις αντισόμενες χώρες, ο δημοκρατικός έλεγχος και σε όλα αυτά τα θέματα είμαστε ε, σκαπανείς η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φυσικά θα πρέπει να εμπλακεί πλήρω και το δικό μα όργανο και οι ευρωβουλευτέ. Θα ήθελα να με διασφαλίσει η Κομισιόν ότι όντω έτσι έχουν τα πράγματα. Δεύτερο, έχουμε 80 μέρε ανοιχτέ για του πολίτε, για του καταναλωτέ, μέρε για την ανάπτυξη για να οργανώσουμε και να ετοιμαστούμε για την υπουργική διάσκεψη. Ίσως θα πρέπει να το είχαμε κάνει ήδη. Αλλά ε, έχουμε και αυτές μερίδες για το διεθνές εμπόριο και μπορούμε να συζητήσουμε μαζί σε αυτά τα πλαίσια το αποτέλεσμα αυτής της διάσκεψης. Η κυρία Μουσκαρντίν για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Μιλήσατε για μείωση της γραφειοκρατίας για διευκόλυνση της μετακίνησης των εμπορευμάτων, γιατί να μην μιλήσουμε με μεγαλύτερη έμφαση για κοινού κανόνες που όλοι πρέπει να σεβαστούμε. Για την καταπολέμηση της πειρατείας και των απομιμήσεων. Δύο λόγια για τις ονομασίες προέλευσης και καταγωγής. Γιατί ε, υπάρχουν χώρες στον ΠΟΕ που είναι χώρες δεύτερη κατηγορία, όπω εμεί. Και το που συναποφάσισε και το Συμβούλιο τι περασμένε μέρε. Ε, 13 χρόνια τώρα δεν γίνεται τίποτα. Κάνουμε μικρά βήματα, αλλά μένουμε στο ίδιο σημείο συνέχεια. Δεν θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Αυτό το κοινοβούλιο από την περασμένη κοινοβουλευτική θητεία είχε ψηφίσει να αλλάξει ο ΠΟΕ να αλλάξει τροχιά. Δεν έγινε τίποτα όμως γιατί πάντα περιμέναμε τα αποτελέσματα της Ντόχα. Τώρα ε, ετοιμαζόμαστε για ένα νέο ραντεβού. Δεν θέλω να περιμένουμε άλλα 13 χρόνια μάταια. Ελπίζουμε τελικά να δοθεί απάντηση και να υπάρξουν κοινοί κανόνες που καθιστούν την ε, αγορά δίκαιη, ελεύθερη και αλληλέγγυα ούτω ώστε να δώσουμε νέα ελπίδα στην ευρωπαϊκή βιομηχανία και να δώσουμε ελπίδα και στις φανάπτυκτες χώρες που ακόμα θεωρούνται ότι είναι στο ίδιο επίπεδο με τις υπερανεπτυγμένες ε, χώρες που έχουν το πλεονέκτημα. Ακριβώς ε, και έχουμε υπόψη μας ας πούμε χώρες όπως η Κίνα που είναι στο ίδιο επίπεδο με τις αφρικανικές χώρες. Δεν γίνεται αυτό. Ένα λεπτό ως Σόλτς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε κύριοι βουλευτέ, όταν αλλάζουν οι παγκόσμιε συνθήκε, θα πρέπει να αλλάζουν και οι συνθήκε του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Και οι διαπραγματεύσει στη Γενέβη έχουν δείξει ότι δεν έχουν υλοποιηθεί οι στόχοι. Η διευκόλυνση του εμπορίου είναι ένα βήμα, αλλά α δούμε τι χρειάζονται και οι αναπτυσσόμενε χώρε. Με τους μικρούς προϋπολογισμούς που έχουν οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν μπορούν να υποχρεωθούν να χρηματοδοτούν έργα υποδομών. Χρειάζονται υποδομές, χρειάζονται νέα λιμάνια, χρειάζονται ε, δυνατότητες για μεγαλύτερες ε, εξαγωγές. Αν δεν τα φροντίσουμε όλα αυτά, η υπουργική διάσκεψη θα αποτύχει. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε υποδομές ε, για το εμπόριο μέσα στη χώρα και να τα υπόψη μας στις διαπραγματεύσεις για τη γεωργία. Αυτό είναι προ όφελο και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο γύρο τη δόχα θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια επικοδομητική πορεία. Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε εμείς για τον υπόλοιπο κόσμο και στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων να εντείνουμε τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου και τον ρόλο τον οποίο παίζει το Κοινοβούλιο σε παγκόσμιο επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, μια ερώτηση. Δέχεστε μια γαλάζια κάρτα από τον κύριο Ρούμπιχ. Κύριε Ρούμπιχ, έχετε το λόγο. Μιλήσατε για τη διευκόλυνση του εμπορίου, κύριε... Ναι, δεν ήταν το μικρόφωνο του κύριου Ρούμπιχ ε, ανοιχτό. Έχω μια ερώτηση λοιπόν κύριε Σόλτς για τη διευκόλυνση του εμπορίου και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βλέπετε να υπάρχει εδώ μια δυνατότητα και για τις δύο πλευρές να επωφεληθούν όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ούτως ώστε να υπάρχουν εμπορικές δραστηριότητες ε, και για τις δύο πλευρές και πώς το συνδέεται αυτό με το γύρο της Ντόχα, ο κύριος Σόλτς. Και βεβαίως βλέπω να υπάρχει ευκαιρία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κύριε Ρουμπιχία, και μάλιστα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να μπορούν να υποφελούνται από την διευκόλυνση για το εμπόριο. Δεν νομίζω ότι αρκεί όμως ε, μόνο αυτό το μέτρο. Και θα έπρεπε να μπορέσουμε εμείς να δώσουμε περισσότερες δυνατότητες στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε με τους επόμενους ομιλητές. Ο κύριος Κασπάρη, μισή λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, λίγες μέρες έχουν μείνει μέχρι την ένατη υπουργική διάσκεψη του ΟΠΟΕ στην Ινδονησία. Εδώ και πολλά χρόνια δεν προχωρεί ο αναπτυξιακός ε, γύρω στην Τόχα. Προσπαθούμε να δώσουμε διάφορες διευκολύνσεις, αλλά δεν έχουμε καταλήξει σε αυτά αποτελέσματα. Οι αριθμοί είναι ξεκάθαροι, δεν νομίζω ότι μπορούμε να το αμφισβητήσουμε, ότι όσο περισσότερο συμμετέχουν οι χώρες στις εμπορικές διαπραγματεύσεις και στην ε, παγκοσμιοποίηση, ε, τόσο, περισσότερο, τόσο περισσότερη ανάπτυξη υπάρχει και το βλέπουμε σε χώρες της Ασίας που έχουν ανοίξει στις διαπραγματεύσεις και έχουν όλο και περισσότερη ανάπτυξη και το βλέπουμε και σε χώρες της Αφρικής που δεν είναι ανοιχτές στις διαπραγματεύσεις και δεν επέρχεται ανάπτυξη. Θα θέλαμε σε αυτή την ένατη υπουργική διάσκεψη να υπάρξει μια βελτίωση. Ίσως κάνουμε ένα μικρό βήμα προς τα μπρος με αυτή, το trade facilitation, αλλά θα πρέπει να περάσουμε και σε άλλους τομείς και νομίζω ότι εκ μέρους ε, της πολιτικής μου ομάδας ε, μπορώ να πω αυτό το οποίο έχουμε επαναλάβει πολλές φορές στο παρελθόν ότι θέλουμε ε, μεγαλύτερη απελευθέρωση και γι' αυτό θα ήθελα να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στους, στον, στην Υπουργική Διάσκεψη. Ευχαριστώ. 1,5 λεπτό κυρία Μακίνες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα, στα, θα ξεκινήσω εκεί που σταμάτησε ο Ντανιέλ Κασπάρη. Πρόσφατα δίνεται μεγαλύτερη σημασία στις διμερείς εμπορικές συμφωνίες και όχι στις παγκόσμιες εμπορικές συμφωνίες στο γύρο της Ντόχα γιατί φαίνεται ότι ε, έχει ξεχαστεί αυτός ο στόχος και γι' αυτό ευχόμαστε κάθε επιτυχία στους διαπραγματευτές. Ο Γενικός Διευθυντής ε, του ΠΟΕ δεν φαίνεται σίγουρος ότι μπορεί να αποσπάσει μια συμφωνία παρόλα αυτά τους ευχόμεθα κάθε επιτυχία. Ε, ε, σταμάτησαν οι διαπραγματεύσει ε, που συνάντησαν ένα τείχο το 2009 λόγω των γεωργικών διαπραγματεύσεων και παραμένει ένα ε, επίμαχο ζήτημα. Ξέρω ότι υπάρχει κάποια πρόοδος, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι έχει επιτευχθεί επαρκής πρόοδος. Και ε, νομίζω ότι ε, υπάρχει η διμερή συμφωνία και της, του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών και θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ προσεκτικά όσον αφορά τις αιτήσει που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον γεωργικό τομέα. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Βάιντερε. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο κόσμος χρειαζόμαστε έναν ισχυρό οργανισμό εμπορίου. Και σε μεγάλο βαθμό οι κανόνες του ΠΟΕ μας έσωσαν από τον προστατευτισμό. Γιατί ιδιαίτερα σε περίοδους κρίσης ε, ο προστατευτισμός ε, ανθεί. Θα πρέπει να συνεχίσουμε λοιπόν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για να αποφύγουμε διακρίσεις στο παγκόσμιο σύστημα εμπορίου. Θέλουμε να διευρύνουμε και να επεκτείνουμε την προσέγγιση της αγοράς, να προασπίσουμε τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, να βελτιώσουμε τη συνεργασία στις, για τη διαμετακόμιση και την τελωνιακή συνεργασία και πιστεύω ότι έτσι θα χαράξουμε το δρόμο για τη Συμφωνία Διευκόλυνση του Εμπορίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μείζον εξαγωγέας υπηρεσιών. Γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό να καταργήσουμε τα εμπόρια ε, για τις επενδύσεις στον τομέα των υπηρεσιών και να το θέσουμε αυτό προτεραιότητα του ΠΟΕ. Επίσης, είναι σημαντικό για όλα τα κράτη-μέλη να συμμορφώνονται με τους κανόνες του ΠΟΕ. Κανένα κράτος μέλος δεν θα πρέπει μονομερός να εφαρμόζει εμπορικές κυρώσεις ή να αλλάζει τις εμπορικές ποσοστώσεις. Γι' αυτό και είναι απαραίτητο να βελτιώσουμε τους μηχανισμούς ελέγχου της συμμόρφωσης με, τις, με τους κανόνες της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου. Σας ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό, κυρία Κιώστιγκερ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Οι διαπραγματεύσει τη ΔΟΧΑ βρίσκονται σε ένα σημείο κοντά στην τελική ευθεία και περιμένουμε να δούμε αν όντω θα μα οδηγήσει, θα μας οδηγήσει η Υπουργική Διάσκεψη ε, στην τελική ευθεία. Ο Γενικό Διευθυντή Αζεβέντο είπε προσφάτω ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στον τελικό στόχο και δεν πρέπει τώρα πια να αποτύχουμε. Η διάσκεψη στο Μπαλί νομίζω ότι ε, θα ε, κάνει τα επόμενα βήματα και θα λυθούν ε, τα ε, ανοιχτά σημεία ε, για τη διευκολύνση στο εμπόριο, για την γεωργία και για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Χρειαζόμαστε ένα αποτέλεσμα από αυτή την Υπουργική Διάσκεψη για να μπορούμε να βελτιώσουμε τη συνολική εικόνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου χρειαζόμαστε ένα κοινό πλαίσιο που θα δίνει τη δυνατότητα στις αναπτυσσόμενες χώρες και στις βιομηχανικές χώρες να αναπτυχθούν ε, σε παρόμοιες συνθήκες εμπορίου. Ένα πολυμερές εμπορικό πλαίσιο ε, θα πρέπει να δοθεί μέσω των διαπραγματεύσεων και ε, είναι προτιμότερο να έχουμε μια πολυμερή συμφωνία και όχι μια σειρά διμερών εμπορικών συμφωνιών η διάσκεψη στον Παλί θα δείξει αν ε, τα κράτη-μέλη έχουν πραγματικά τη βούληση να στηρίξουν ένα ισχυρό ΠΟΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα στηρίξει αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κέλεμ, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε. Ίσως ε, θα πρέπει να ξεχνούμε ότι μια συνολική αναπτυξιακή ατζέντα της Δόχα θα αυξήσει τις παγκόσμιες εξαγωγές για πάνω από 300 δισεκατομμύρια ευρώ, για πάνω από 2% δηλαδή. Ιδιαίτερα τη σήμερα ημέρα θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εφαρμόσουμε πιο αποφασιστικά και σωστά ένα εμπορικό σύστημα χωρίς, διακριτικές, χωρίς διακρίσεις με κοινέ αξίες και υιοθέτηση παγκόσμιων προτύπων και προδιαγραφών. Κάτι τέτοιο όμως προϋποθέτει διαρθρωτική μεταρρυθμίση παγκόσμιας οργάνωσης εμπορίου και φυσικά να γίνουν δεκτές αυτές οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε συγκεκριμένες προτεραιότητες. Πρώτον, να μειώσουμε τους φραγμούς στο εμπόριο και τις επενδύσεις, ιδιαίτερα στον τομέα των υπηρεσιών, ιδιαίτερα τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών, ηλεκτρονικό εμπόριο και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Δεύτερον, ιδιαίτερη έμφαση στη, στο ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο διεθνέ εμπόριο, δηλαδή απλούστευση των κανόνων. Και τρίτον, να βοηθήσουμε τις ε, λιγότερο ανεπτυγμένε χώρες. Κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να στενιστούμε την πρωτοβουλία Everything ε, But Arms, που προσφέρει 100% ε, φορολόγητες και χωρίς ποσοστώσεις προσβάσεις στην αγορά για τις λιγότερο ανεπτυσσόμενες χώρες για την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλό θα ήταν να μειώσουμε και τις ε, γεωργικές επιχορηγήσεις κατά 80% γιατί αυτές είναι που στρεβλώνουν το εμπόριο. Σας ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στη διαδικασία Catch the Eye. Ο κύριος Ρούμπιχ είναι ο πρώτος ομιλητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βρισκόμαστε ενώπιον των πλέον σημαντικών αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν στους επόμενους μήνες. Θέλουμε να ξεπεράσουμε την κρίση στην Ευρώπη και να δημιουργήσουμε τις γενικότερες συνθήκες, ούτω ώστε η οικονομία μας ε, να μπορέσει να προχωρήσει σε ένα σίγουρο μέλλον για την Ευρώπη. Γι' αυτό το βασικό ερώτημα είναι πώς μπορούμε να τα καταφέρουμε σε διεθνές επίπεδο, ώστε να προχωρήσουν οι πολυμερείς ε, συμφωνίες ή αν θα μείνουμε στην τωρινή κατάσταση χωρίς καμία πρόοδο. Αν δεν γίνει τίποτα θα τεθεί ένα άδοξο τέλος στο γύρο της Δόχα. Τώρα έχουμε τη δυνατότητα το Δεκέμβριο να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία της Δόχα αυτά τα οποία έχουν γίνει μέχρι τώρα θα πρέπει να συμπληρωθούν, να ολοκληρωθούν γιατί ακόμη και σε περίπτωση που αποτύχουν αυτές οι προσπάθειες θα χρειαστεί μια ατζέντα για μετά την Τόχα. Ευχαριστώ. Η κυρία Κέλλερ, τελευταία ομιλητρία. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Οι Ηνωμένε Πολιτείε πάντοτε μιλούν υπέρ των πολύπλευρων συμφωνιών, αλλά ε, από το 2007 το υπονομεύουν με διμερείς περιφερειακές ή πολυμερείς συμφωνίες. Χρειαζόμαστε πραγματική δέσμευση των πολυμερών συμφωνιών και γι' αυτό χρειάζεται μια διαρθρωτική μεταρρύθμιση του ΠΟΕ για να υπάρχει ένα δίκαιο σύστημα εμπορίου που θα βασίζεται σε ισότιμους κανόνες που θα λαμβάνουν υπόψη τι παγκόσμιες προκλήσει όπως την αλλαγή του κλίματος, την ένδυα, τον κοινωνικό αποκλεισμό, την ανισότητα των φύλων και την μετανάστευση να έχει ιδιαίτερη σημασία οι αναπτυσσόμενες χώρες και ιδίως οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες ε, να συμμετάσχουν πλήρως σε αυτές τις διαπραγματεύσεις της ένατης υπουργικής διάσκεψης στο Μπαλί. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να φροντίσει να συμμετάσχουν και αυτές οι χώρες, ιδίως ε, για την εξασφάλιση της πρόσβασης στην αγορά χωρίς δασμούς και χωρίς ποσοστώσεις, καλύτερες λύσεις για το βαμβάκι και ε, καλύτερη αντιμετώπιση της εξαίρεσεις για τις υπηρεσίες. Θα πρέπει να συμμετάσχουν ενεργά και οι λιγότερο ενεπτυγμένες χώρες για να επιτύχει ο γύρος της ΔΟΧ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές και δίνω το λόγο στην κυρία Ρέντινγκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. λέει με τους συνεργάτες μου σημείωσα τις σημαντικές παρεμβάσεις των Ευρωβουλευτών και θα τις λάβουμε υπόψη γιατί οι ευρωβουλευτές ούτως ή άλλως θα είναι τμήμα της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας και θα είναι παρόντες στα τεκτενόμενα και ούτως ή άλλως κατά τη διάρκεια της διάσκεψης και με τη διάσκεψη θα μπορούμε να ανταλλάξουμε περαιτέρω απόψεις. Μια ερώτηση έγινε για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε διαφορά την επικύρωση. Μεταξύ των αποφάσεων του ΠΟΕ που θα ληφθούν στη διάσκεψη του Μπαλί, μόνο λίγες θα έχουν ε, νομική ισχύ. Παραδείγματο χάρη άρθρο 218 κάθετος 9 της συνθήκης. Ε, αυτό λέει. Ε, ασφάλεια, μηχανισμός παρακολούθησης για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Μόνο, για αυτές μόνο αποφάσεις του Συμβουλίου προβλέπονται. Μία διευκόλυνση του εμπορίου θα ολοκληρωθεί ως ε, ενοποιημένη νέα συμφωνία του ΠΟΕ και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ε, με εξαίρεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, θα παρακολουθήσουν τις εσωτερικές διαδικασίες με βάση το άρθρο 2.18 κάθετος 6. Και αυτό θα γίνει έξι μήνες μετά την ε, διάσκεψη του Μπαλί. Ευχαριστώ κύριε πίτροπε. Έχω τρεις προτάσεις ε, για ψηφίσματα από τους πράσινους, από την ΚΟΕ και από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Κλείνουμε εδώ τη συζήτηση και θα ψηφίσουμε αύριο στις 12 η ώρα το σημείο αυτό. Τώρα κυρίες και κύριοι, πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάδαξης που είναι σημείο του κυρίου Μαρινέσκου για τα ευρωπαϊκά συστήματα δορυφορικής πλοήγησης. Θα ήθελα καταρχήν να δώσω το λόγο στον κύριο Μαρινέσκου για τέσσερα λεπτά.